ο επισκέπτης έχει μάλλον κάποια προσωπικά προβλήματα, θα ασχοληθούμε μαζί του. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου εχθές ενέκρινε την έκθεση για τη Συμφωνία για το Κλίμα του Παρισιού. Έτσι, ε, πληρούνται και οι τυπικές προϋποθέσεις έτσι ώστε σήμερα η Ολομέλεια να ψηφίσει την έκθεση που θα μας παρουσιάσει ο συνάδελφος Λαβία. Πρόκειται για μια ιστορική ψηφοφορία, διότι με την έγκριση του παρόντος κειμένου κάνουμε το τελευταίο πολιτικό βήμα στο δρόμο προς την κύρωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Με την ψηφοφορία μας αυτή ανοίγει πλέον ο δρόμος έτσι ώστε η συνολική συμφωνία να μπορέσει να ξεπεράσει τις προβλεπόμενες ε, οριακές τιμές και το κατόφλι για να τεθεί σε ισχύ. Δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος από την έγκριση της συμφωνίας το Δεκέμβριο του 2015 και αυτό το αποτέλεσμα θα ήταν πραγματικά ε, συγκλονιστικό και μάλιστα πριν τη διάσκεψη του Μαρακές COP22. Άρα έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτόν τον τρόπο θα επεδείκνει ηγετικό ρόλο. Για να συγκρίνουμε μόνο, από τη στιγμή που εγκρίθηκε το πρωτόκολλο του Κιώτο μέχρι να τεθεί σε ισχύ, ε, παρέλθαν 8 έτη. Και τώρα βρισκόμαστε σχεδόν 9 μήνες μετά τη διάσκεψη ε, των Παρισίων. Γι' αυτό έχω την ιδιαίτερη χαρά που συμφωνήσατε αγαπητοί συνάδελφοι με την πρότασή μου να το γιορτάσουμε αυτό σε μια πανηγυρική συνεδρίαση όπως αρμόζει. Και είναι πολύ μεγάλη τιμή που νιώθουμε που ο Γενικός Γραμματέας των Ομένων Εθνών, ε, κύριος Μπαν Κιμούν, έχει έρθει στην Ολομέλειά μας. Είστε χωρίς καμιά αμφιβολία ένας από τους πιο μεγάλους αρχιτέκτονες αυτής της ιστορικής συμφωνίας. Και σας καλωσορίζουμε θερμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τιμούμε και ξέρουμε το ρόλο που έχετε διδραματίσει στην κατεύθυνση αυτή. Θέλουμε σήμερα να ευχαριστήσουμε και τη Γαλλική Δημοκρατία που φιλοξένησε την COP21, τη διάσκεψη αυτή και κατέβαλε τεράστιες πολιτικές προσπάθειες έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα αυτή η συμφωνία. Και χαίρομαι πάρα πολύ που η Προεδρεύουσα της διάσκεψης COP21 παρευρίσκεται Κυρία Υπουργέ, ε, κυρία Ρουαγιάλ, θα ήθελα στο πρόσωπό σας να ευχαριστήσω το σύνολο ε, της γαλλικής κυβέρνησης για τις εξαιρετικές και καταπληκτικές προσπάθειες θα μας απευθύνει το λόγο και θα μας θυμίσει ο Γενικός Γραμματέας του ΕΕ, κ. Μπαν και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους προέδρους των πολιτικών ομάδων και μετά θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Κύριε Γενική Γραμματέα, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Εξοχότατε, κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Μάρτιν Σούλτ. Εξοχότατε, κύριε Ζωάν Κλοντ Ιούνκερ, Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εξοχότατε, κύριε Κόρτσοκ, Πρόεδρε και ε, ε, Υπουργέ ε, Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Προεδρέμοντα του κοπη 22 αξιότιμη κύριε Τσεύκοβιτ, αντιπρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπεύθυνη για την κλιματική αλλαγή, αξιότιμη κύριε Άρια Κανιέτε, Επίτροπε για το περιβάλλον, αξιότιμη κύριε Λαβία, πρόεδρε της Επιτροπή περιβάλλοντο Υγεία και Προστασία του Καταναλωτή, αξιότιμη μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμη Υπουργή κυρίε και κύριοι. Οτελεί για μένα μεγάλη τιμή ως Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να απευθυνθώ στα αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ για αυτή την τιμή που μα κάνετε. Κατάφερα να αλλάξω το πρόγραμμα των ε, ταξιδίων μου για να έχω την ευκαιρία να παρευρεθώ σε αυτήν την πανηγυρική συνεδρίαση μετά την ε, πρόσκληση του κυρίου Σούλτς. Σήμερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επικυρώσει τη Διεθνή Συμφωνία για την Κλιματική Αλλαγή. Εκτιμώ την συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στον τομέα της κλιματικής αλλαγής. Μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις του καιρών μας. Ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχετε αποδείξει ότι αντιμετωπίζετε το ζήτημα αυτό με τη σοβαρότητα που του αρμόζει, ότι αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι, αλλά ταυτόχρονα καταλαβαίνετε ότι και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μπορεί να οδηγήσει σε μια βιώσιμη ε, οικονομία και βελτίωση των ε, κοινωνικών συνθήκων. Κατά την διάρκεια των διαπραγματεύσεων είχατε μια επικοδομητική στάση, έχετε δημιουργήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση το, το, ε, το πράσινο ταμείο. Με πολλούς λοιπόν τρόπους έχετε αποδείξει την ε, προσήλωσή σας στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σήμερα σας ζητώ να αξιοποιήσετε αυτά τα προηγούμενα βήματα και να κάνετε ακόμα ένα βήμα να προχωρήσετε στην επικύρωση της ε, Συμφωνίας για την Κλιματική Αλλαγή. Κάτι που θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη της να ε, καταθέσουν το έγγραφο επικύρωσης ε, στο γραμματεία του ΟΗΕ. Είναι εντυπωσιακή οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία αυτή η συμφωνία είναι ακόμα πιο σημαντική και ακόμα εντυπωσιακότερη ακριβώ επειδή αντιμετωπίζει ένα από τα σημαντικότερα θέματα που ε, προβληματίζουν τον κόσμο σήμερα. Τα τελευταίους μήνες έχουμε ε, σημειώσει ε, μεγάλη πολιτική βούληση να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία. Τον Σεπτέμβριο, στις 21 Σεπτεμβρίου, στον ΟΗΕ Πολλέ χώρε εκπροσωπήθηκαν σε μια συναντήση υψηλού επίπεδου την οποία διοργάνωσε και στην οποία κατατέθηκαν τα έγγραφα επικύρωση από δύο από τι σημαντικότερε χώρε, από εκείνε που ε, εκπέμπουν ε, το μεγαλύτερο ποσοστό ε, αερίων του θερμοκηπίου, τι ΗΠΑ και την Κίνα. Εάν σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση επικυρώσει, σημαίνει ότι θα έχουμε ξεπεράσει το κατόφλι, θα έχουμε 62 χώρες που θα έχουν επικυρώσει τη Συμφωνία του Παρισίου. Ξεωτήμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, αντιλαμβάνομαι ότι η διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ξεχωριστή. Θέλω να σημειώσω την απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος ε, η οποία ελέγχθη στο Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουν με εγωριέ διαδικασίε, με fast track στην επικύρωση τη συνθήκη του Παρισιού. Σα ζητώ να δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη συγκατάθεσή του σε αυτή την ταχεία διαδικασία. Έτσι ώστε γρήγορα να ξεπεράσουμε το ελάχιστο κατόφλι που χρειάζεται, έχετε τη δυνατότητα να γράψετε ιστορία, να δώσετε τον, τη δυνατότητα στον κόσμο να ελπίζει σε ένα καλύτερο μέλλον. Έτσι ώστε η Συμφωνία του Παρισίου να επικυρωθεί και να τεθεί σε εφαρμογή σε χρόνο ρεκόρ. Αυτή η γρήγορη ε, θέση σε ισχύ θα αποδείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προσιλωμένη στη διεθνή συνεργασία, η οποία εξάλλου βρίσκεται στην καρδιά της ταυτότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να πάμε προ μια κατεύθυνση μια οικονομία, η οποία θα έχει χαμηλέ εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα να καταπολεμήσουμε την αύξηση τη ε, θερμοκρασία και να επιτύχουμε το στόχο για αύξηση τη θερμοκρασία αρκετά κάτω από του δύο βαθμού Κελσίου. Επίση πρέπει να βοηθήσουμε εκείνε τι χώρε που πλήττονται από την κλιματική αλλαγή να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο. Στο όνομα του ανθρωπισμού, στο όνομα των επόμενων γενεών, σας ζητώ να εγκρίνετε την ταχεία επικύρωση της Συμφωνίας του Παρισίου για την κλιματική αλλαγή. Ξεότιμη κύριε Πρόεδρε, εξοχότατη μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να έχετε τη δυνατότητα να αναλάβετε ιστορική δράση. Σε μια περίοδο όπου οι διαιρέσεις και οι διχασμοί αυξάνονται, έχουμε τη δυνατότητα, έχετε τη δυνατότητα να αποδείξετε ότι είστε ενωμένοι και ότι ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε ένα, ένα πιο δίκαιο και πιο βιώσιμο μέλλον. Ας αδράξουμε λοιπόν αυτή την ευκαιρία και ας ανταποκριθούμε στις αξίες και στους στόχους των οργανισμών που υπηρετούμε. Ξεκινούμε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξεκινούμε Υπουργοί, ξεχότατοι. Όπως γνωρίζετε, η θητεία μου ως Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ τελειώνει φέτος. Ήταν για μένα πολύ μεγάλη τιμή να υπηρετήσω αυτόν τον πολύτιμο διεθνή οργανισμό και να συνεργαστώ στο πλαίσιο αυτό με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιο συγκεκριμένα. Θα ήθελα λοιπόν ε, με την ευκαιρία που μου δίνετε σήμερα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για την υποστήριξη που μου παρήχατε τα τελευταία δέκα χρόνια και προσωπικά και προς τον Οργανισμό Ενωπαίνων Εθνών. Είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ηγείται στους τομείς ε, που ενδιαφέρουν τα Ηνωμένα Έθνη, δηλαδή στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο περιβάλλον, στην, στα κοινωνικά θέματα. Ας συνεχίσουμε λοιπόν να αγωνιζόμαστε μαζί για να γίνει ο κόσμος καλύτερος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Γραμματεύ. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί τώρα η διαδικασία της ψηφοφορίας. Καταρχάς, να σας εξηγήσω σύντομα τη διαδικασία. Θα μιλήσουν πρώτα οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων. Θα κάνουν μια σύντομη δήλωση, ο καθένας εξ ονόματος της ομάδας του. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Και τέλος, όπως είπαμε προηγουμένως, θα δώσω το λόγο βάσει του κανονισμού μας τον εισηγητή και πρόεδρο της Επιτροπή Περιβάλλοντος, κ. Τζοβάνι Λαβία. Μετά θα ψηφίσουμε ονομαστικά. Σε περίπτωση έγκρισης, ολοκληρώνεται η διαδικασία συνένεσης του Κοινοβουλίου τυπικά και θα υπογράψω την διαβαστική επιστολή προς τον πρόεδρο, του Συμβουλίου, τον πρόεδρο μάλλον του Συμβουλίου. Και θα υπογράψει ο κύριος Γενικός, η κύριε Υπουργός Ροαγιάλ και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με αυτή τη διαβαστική επιστολή μπορεί να κάνει τις υπόλοιπες ενέργειες στο Συμβούλιο για την κατάθεση του εγγράφου στη Νέα Υόρκη και επιτυχάνεται το κατόφλι 55% ε, που χρειάζεται και μάλιστα το υπερβαίνουμε έτσι ώστε να τεθεί σε ισχύ η Παγκόσμια Συμφωνία για το Κλίμα. Μετά την ψηφοφορία θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, του Συμβουλίου, την κυρία Ρουαγιάλ, τον Γενικό Γραμματέα και τον κύριο Λαβία να έρθουν για να υπογράψουμε. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα το λόγο έχει τώρα ο Πρόεδρος κύριος Βέμπερ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέα, καταρχάς καλώς ορίσατε θερμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας πω ότι και εμείς σας ευχαριστούμε για το έργο σας, για ό,τι κάνετε για τον κόσμο τελευταία δεκαετία και την εταιρική σχέση με την Ευρώπη. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κλιματική αλλαγή είναι ίσως το υπαριθμό ένα καθήκον της δικής μας γενιάς πολιτικών. Γι' αυτό και η σημερινή μέρα είναι όντω ιστορική. Και οι Ευρωπαίοι μπορούν να είναι περήφανοι διότι εμείς ε, ανέκαθεν ήμασταν η ηγέτιδα Ήπειρος για να ε, ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Χωρί την ηγετική πρωταγωνιστική στάση τη Ευρώπη δεν θα μπορούσε να έχει υπογραφεί. Και μάλιστα έπαιξε μεγάλο ρόλο το γεγονό ότι ήμασταν ενωμένοι με μια φωνή απέναντι σε παγκόσμια θέματα. Και δείχνει αυτό πραγματικά τι μπορούμε να κάνουμε εμεί οι Ευρωπαίοι όταν είμαστε ενωμένοι. Μετά την υπογραφή, τώρα όμω χρειάζεται και δράση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή οι δεσμεύσει και οι υποσχέσει θα πρέπει να υλοποιηθούν. Εξ ονόματο τη δική μου ομάδα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι κατά την άποψή μα τα παγκόσμια προβλήματα χρειάζονται παγκόσμιε λύσει. Παρά το λαϊκισμό που σηκώνει κεφάλι παγκοσμίω, εμείς δείχνουμε ότι τα παγκόσμια προβλήματα μπορούμε να τα λύνουμε από κοινού. Πολλά προβλήματα, πολλές ανησυχίες και μελήματα είναι κοινά. Ε, σήμερα όμως είναι μια μέρα αισιοδοξία. Σήμερα δείχνουμε τι μπορούμε να λύσουμε. Γι' αυτό είναι ιστορική και καλή η σημερινή ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Από τους σοσιαλδημοκράτες το λόγο έχει ο Πρόεδρος Πιτέλα. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη ε, κυρίες και κύριοι, η κυρία Ροαγιάλ σε κολέρο για άλλα. Εξοχότατε, Μπάνκι σας ευχαριστώ για την ε, δεκαετή σας προσήλωση ε, στο θέμα αυτό και που την αισθενιζόμαστε κι εμείς και η Ευρώπη του σήμερα είναι πραγματικά η Ευρώπη που επιθυμούμε. Όχι η Ευρώπη που ομφαλοσκοπεί, που είναι κλειστή στον εαυτό τη, αλλά μια Ευρώπη ανοιχτή στον κόσμο και που υλοποιεί την πρωταρχική της αποστολή, που είναι αυτή να μεριμνήσει για τους ανθρώπους ε, και για τη γη η Ευρώπη στην υπηρεσία μιας καλύτερης ζωής και όχι ένα συνοθήλευμα νομικών γραναζιών. Σήμερα γράφουμε ιστορία, κύριε Βέμπερ. Δίκιο έχετε. Αλλά θα πρέπει να αναλάβουμε και άλλα καθήκοντα, να μεταφέρουμε τη θεωρία, αυτά που έχουμε συμφωνήσει και γράψει στην πράξη και να έχουμε και πιο φιλόδοξες ε, αποστολές. Γιατί η Γη, ο πλανήτης μας ε, που εμφανίστηκε μερικά ε, δισεκατομμύρια πριν και που ο άνθρωπος έχει μόνο πολύ λίγο τμήμα αυτής της ιστορίας. Δεν ανήκει σε εμά η Γη. Θα πρέπει να τη διαφυλάξουμε, να τη φροντίσουμε και να την διαβιβάσουμε στα παιδιά μας. Ευχαριστώ από τους συντηρητικού και μεταρρυθμιστές. Το λόγο έχει βουλευτής ο κύριος Μέσσερσμιτ. Ευχαριστώ. Δεν είναι σαφές ότι η συμφωνία της περισμένης Παρασκευής ε, θα απέβαινε στην κύρωση της συμφωνίας. Όπως αναγνωρίστηκε, τώρα το μονοπάτι έχει ανοίξει για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει και την επίσημη συνένεση όπως προβλέπει η συνθήκη. Η υιοθέτηση της συμφωνίας αυτής μετά τις ε, δηλώσεις της COP21 για τις ε, 187 ε, ε, μέρη και τις ε, καθορισμένες υποσχέσεις και εθνικές δεσμεύσεις θα οδηγηθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις ΗΠΑ και άλλες 60 χώρες μέλη που κατέθεσαν τα, τις κυρώσεις τους να οδηγηθούμε ώστε να γίνει δεσμευτική μέχρι τέλη του έτους Συμφωνία των Παρισίων η συμφωνία αυτή είναι σημαντική για όλους, ε, για τους επενδυτές, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τους πολιτικούς ηθήνοντες, γιατί πραγματικά 189 ε, ήταν τα εθνικά ε, σχέδια κλιματικών αλλαγών που κατατέθηκαν και αυτό δείχνει πόσο σφαιρικό είναι αυτό το έργο. Και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί αυτή η κυρώση και να δούμε πώς οι εθνικές κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσουν τις, υποθε... υποσχέσεις που έχουν πραγματοποιήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Από την Ενωτική Αριστερά το λόγο έχει η πρόεδρος της ομάδας, κυρία Τσίμερ. Κύριε Φερχόφστατ, ξέχασα τους φιλελευθέρους. Το λόγο έχει η κυρία Φερχόφστατ. Και στη συνέχεια η κυρία Τσίμερ. Παρακαλώ κύριε Φερχόφστατ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενική Γραμματέα, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή τη δεκαετία τη δεκαετή θητεία σας και κύριε Πρόεδρε ε, χαίρομαι που ήρθατε, που βρήκατε το δρόμο προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μάλιστα ε, έχετε λάβει και πρόσκληση να έρθετε στην ε, Επιτροπή εμείς. Γνωρίζετε πια το δρόμο. Αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι η Συμφωνία των Παρισίων ε, της COP21 έχει ιστορική σημασία και κατά τη γνώμη μου είναι τόσο ιστορική όπως και η Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948. Όπως και το 1948, όπως και τότε, σήμερα η COP21 αποδεικνύει ότι η πολυμερής προσέγγιση λειτουργεί και ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση για τον πλανήτη δεν είναι ουτοπία, δεν είναι όνειρο όπως ισχυρίζονται μερικοί. Και επίσης αποδεικνύει ότι η Ευρώπη μπορεί να πρωτοστατήσει και να οδηγήσει τον κόσμο προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι εν τη ενός ισχύς από κοινού είμαστε ισχυρότεροι. Τι δραματική διαφορά σε σχέση με την τραγωδία που εκτιλήσατε στο Χαλέπι, όπου άμαχος πληθυσμός χάνει τη ζωή του, βομβαρδίζονται νοσοκομεία, ε, έχουμε φτάσει σε αντιέξοδο σχέσεις ε, Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών και μάλιστα ε, απροθυμία του ενός, βάναυση και αμήλικτη αποφασιστικότητα και πυγμή του άλλου. Αυτή είναι η μεταπολεμική <laughs> λογική του Συμβουλίου Ασφαλείας. Γι' αυτό η COP21, η Συμφωνία των Παρισίων, αποδεικνύει ακριβώ το αντίθετο, ότι η παγκόσμια κοινότητα και η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναλάβουν τι ευθύνε του και ότι η πολυμερή προσέγγιση είναι ο ακολουθητέο δρόμο για τι επερχόμενε γενιέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φερχόφστατ και ζητώ και πάλι συγγνώμη. Παρακαλώ να με συμπαθάτε. Τώρα όμως έχει το λόγο εξ ονόμα της Ενωτική Αριστεράς η πρόεδρο κυρία Τσίμερ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, είμαι πρόθυμος, πρόθυμη στο μέλλον να μιλώ και πρώτη εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Μπορούμε να το εγκαινιάσουμε και αυτό, δεν έχω πρόβλημα. Ε, αξιότιμη κύριε Μπανκιμού, θα ήθελα και εγώ εξ ονόματο τη ομάδα μου να σας καλωσορίσω εγκάρδια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ μεγάλη τιμή για μα. Η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής είναι παγκόσμια πρόκληση και σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Δημιουργήθηκε ένα δεσμευτικό πλαίσιο για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Πλην όμω και θέλω να το πω και αυτό, η σημερινή απόφαση και η σημερινή πράξη για μας είναι αφετηρία. Δεν μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς. Θα πρέπει να προχωρήσουμε, να δούμε με ποιο τρόπο ζούμε, με ποιο τρόπο παράγουμε, με ποιο τρόπο καταναλώνουμε. Αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει γενικά ο καπιταλισμός. Ας συμφωνήσουμε λοιπόν πώς θέλουμε παγκόσμια να ζούμε όλοι μαζί, να τα σε αυτή την ευθύνη δεν είναι μόνο το περιβάλλον, είναι και η κοινωνική ζωή και είναι και η συνύπαρξη ε, με τα ζώα και ε, με τη φύση γενικότερα και πώς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό βιώσιμα και αηφόρα. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεδομένοι. Έχουν συμφωνηθεί για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, αλλά δεν αρκούν. Τέσσερα ευρώ τον τόνο δεν αρκεί ως τιμή για την εμπορία εκπομπών. Δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα για τα καυσαέρια. Ε, ούτε είναι αυτό σύγχρονο χάρτη. Αυτό θέλουμε ε, λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε και το χρωστάμε στα παιδιά μας. Από τους Πρασίνους το λόγο έχει η Πρόεδρος κυρία Χάρμς. Εξαιρετούμε κύριε Γενική Γραμματέα Μπανκιμούν. Κιμούν. Ακριβώς επειδή πιστεύω ότι σπαράζει και η δική σας καριά κάθε μέρα, κοιτάζοντας τη Συρία, θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσά και στα Ηνωμένα Έθνη και να σας συγχαρώ για κάτι το οποίο τουλάχιστον επέτυχε. Γιατί για τη συμφωνία του Παρισίου μπορούμε να το πούμε πλέον και για τη διαδικασία κύρωσής της. Και πραγματικά είμαι ακράδαντα πεπισμένη ότι η συμφωνία αυτή θα αποτελέσει κάτι σημαντικό και για τη διεθνή προστασία του κλίματος, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό για τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, το οποίο υγείστε μέχρι τα τέλη του έτους. Θα σας ευχόμουν να επιτύχετε κάτι και εκεί απέναντι σε αυτή τη φρίκη που βλέπουμε στη Συρία και στο Χαλέπι. Από την κυρία Ροαγιάλ, εμείς τι περιμένουμε, η πράσινη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορώ να το πω αυτό, περιμένουμε το Συμβούλιο να μην κυρώσει μόνο και να μην δείξει ικανότητα για λήψη αποφάσεων, αλλά και ικανότητα για φιλόδοξη δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όλες τις τεχνολογίες για να παράγει διαφορετικά. Μπορούμε να, παράγουμε διαφορετικά ενέργεια, να οργανώσουμε διαφορετικά τις μεταφορές μας. Αλλά επιτέλους ε, θα πρέπει να κάνουμε άλματα και όχι διστακτικά βήματάκια. Ε, η ε, συνέπεια που αποδεικνύεται σήμερα εδώ και επιδεικνύεται θα πρέπει να επιδειχθεί και στο μέλλον και από τους ηγέτες μας. Τι κάνουμε εμείς στην Ευρώπη και το πώς παράγουμε στα βιομηχανικά κράτη αυτού του κόσμου. Αυτό έχει αποφασιστική σημασία για το μέλλον των ανθρώπων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι μόνο σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Το θέμα ε, βέβαια, της προσφυγιά δεν πρόκειται να το συζητήσουμε εδώ, αλλά η Συμφωνία για το Κλίμα είναι τεράστια πρόκληση και οι Ευρωπαίοι τα τελευταία χρόνια ε, ήταν φιδουλοί στη φιλοδοξία. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. E Από την ομάδα e FTT το λόγο έχει ο βουλευτής κύριος Πεντιτσίνη. Grazie, Ευχαριστώ. Και εμεί ε, ε, νιώθουμε ικανοποιημένοι από την κύρωση τη Συμφωνία των Παρισίων εκ μέρου Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια δεν αρκεί η κύρωση. Δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε αυτό το πρώτο βήμα, αλλά αντίθετα να πολλαπλασιάσουμε τις δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τις βασικές προκλήσεις στο μέλλον. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα λόγια του Φικέρης. Αν δεν αντιστρέψουμε τις στάσεις ε, την επόμενη πενταετία θα προκαλέσουμε τεράστια ανθρώπινη οδύνη. Κάτι που είναι απαράδεκτο. Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το αλόκοτο και παράλογο μοντέλο του παρελθόντος που στηρίζεται σε μια ξέφραγη ανάπτυξη σαν να είχαμε ανεξάντλητους πόρους. Θα πρέπει να αντικαταστήσουμε αυτό το μοντέλο με ένα μοντέλο ισορροπίας. Ο 9χρονος γιος μου μου είπε πριν από λίγε μέρες ότι αν ψηλώνουμε συνεχώς θα χτυπήσουμε το κεφάλι μας στο ταβάνι. Αυτό θα πρέπει να κάνουμε, να δούμε τον κόσμο από τα μάτια ενός παιδιού, γιατί στα παιδιά αυτά θα αφήσουμε ως παρακαταθήκη τη γη μας. Από την ομάδα ΕΝΕΦ, ο πρόεδρος Δεκράφ έχει το λόγο. Τι θα κάνουμε για την κλιματική αλλαγή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία σχέση και δεν θα πρέπει να κυρώνει αυτή τη συμφωνία του Παρισιού. Και πάλι βλέπω χαρούμενα πρόσωπα εδώ, γιατί υποτίθεται ότι έχουμε ιστορικό ορόσημο σήμερα. Τα κατανοώ όλα αυτά ως ε, προφανή επιρροή σε αυτή τη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ε, μονομερώς ε, μεροληπτικές εις βάρος των αναπτυσσόμενων χωρών συμφωνίες. Τα κράτη-μέλη έχουν να υπομισθούν διάφορα βάρη. Χαίρεται εδώ η ελίτ, γελάει και τρίβει τα χέρια της γιατί θα υποφεληθεί από τα σχέδια αυτά για το περιβάλλον. Αλλά οι ε, σκληρά εργαζόμενοι πολίτες θα πληρώσουν πιο ακριβά το αυτοκίνητό του τη θέρμανση, το ρεύμα, ό,τι άλλο θέλετε. Έσχος είναι αυτά τα πράγματα. Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρώνει αυτό το γεγονός και εγώ βλέπω μόνο ένα φωτεινό σημείο. Δεν είναι δεσμευτικό για τα κράτη-μέλη. Ε, κατά το δοκούν μπορούν να τα κυρώσουν, να τα εφαρμόσουν όπως θέλουν. Και αυτό είναι το θετικό. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Μπαλτσό, μη εγγεγραμμένος βουλευτής. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. nagyon θα ήθελα να πω ε, ότι σήμερα υποτίθεται ότι πανηγυρίζουμε εδώ και ε, εορτάζουμε. Μα ακούτε τώρα, ε, θα πρέπει να υπογράψουμε ένα επίσημο έγγραφο. Να επανέλθω, να αρχίσω γιατί είχαμε ένα τεχνικό πρόβλημα ξανά. Έλεγα λοιπόν ότι τώρα μακούτε, ακούτε. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα στη διερμηνία. Παρακαλώ. Ωραία. Αρχίστε και πάλι από την αρχή, λέει ο Πρόεδρος. Ωραία. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κύριε Γενικέ Γραμματέα. Βλέπουμε στην ενημερήσια διάταξη εδώ να λέει πανηγυρική συνεδρίαση. Τι πανηγυρική. Εδώ είναι πολύ σημαντικά τα ζητήματα ουσίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να επικυρώσει αυτή τη συμφωνία και πολλά κράτη το έχουν πράξει και μεταξύ αυτών και η Ουγγαρία. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα ε, για να τεθεί σε ισχύ αυτή η συμφωνία. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο κατά της κλιματικής αλλαγής, έχουν στόχους φιλόδοξους, διατυπώσει και συμφωνήσει. Ωραία. Τώρα όμως αν το θέμα είναι να μπούμε σε μια κούρσα ποιο έχει πιο φιλόδοξου στόχου, επιτρέψτε μου να κάνω τι εξή παρατηρήσει. Εμεί έχουμε ευθύνη ε, για τους Ευρωπαίους πολίτες και για την ευρωπαϊκή οικονομία. Και τα βήματα που κάνουμε είναι και πιο ακραία και ριζικά. Πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι η Ευρώπη είναι υπεύθυνη μόνο για το 10% της εκπομπής ρήπων. Και αυτό που μας ενδιαφέρει ε, δεν είναι μείωση των ρήπων, αλλά ε, με την κατάσταση ουσιαστικά των ρήπων, εξαγωγή των ρήπων. Ε, θα πρέπει να παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή οικονομία και να μην σηκώνονται να φεύγουν οι επιχειρήσεις. Αυτό που έχει σημασία είναι να είναι νομικά δεσμευτική μια συμφωνία, λέτε, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να τα εφαρμόσει όλα αυτά. Ε, δεν είναι δυνατόν οι Ηνωμένε Πολιτείε, που είναι μια από τι μεγαλύτερε οικονομίε αυτή τη γη, να ε, ε, ε, εκπέμπουν τα περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου και να ρηπαίνουν περισσότερο και να εξυπηρετούν μόνο τα αμερικανικά συμφέροντα. Θα πρέπει ο καθένας να καταλάβει ποιος είναι ο ρόλος του και να τον επομιστεί. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο έχει ο πρόεδρος, ο κύριος Γιούνκερ. Monsieur le Président, Monsieur... κύριε Γενικά Γραμματέα, κύριε Πρόεδρε, σήμερα αποδεικνύουμε ότι είμαστε ικανοί όταν συνεργαζόμαστε να ε, καταφέρνουμε μεγάλα επιτεύγματα. Η συμφωνία του Παρισίου δεν έπεσε από τον ουρανό. Χρειάστηκε να συνεισφέρουν ε, πολλοί από εμάς. Θα ήθελα να συγχαρώ τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, τον κύριο Ολόντ, τον κύριο Λογόν Φαμπιούς και την κυρία Ρουαλιάλ. Γιατί επέδειξαν ε, προσήλωση και εργάστηκαν σκληρά έτσι ώστε τελικά να φτάσουμε σήμερα να μπορούμε να επικυρώνεται αυτή η συμφωνία. Μέσα σε ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο είχα δηλώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να επικυρώσει οποιαδήποτε συμφωνία για το κλίμα, αλλά παρά μόνο μια συμφωνία η οποία θα ήταν φιλόδοξη και ουσιαστική. Και τα καταφέραμε. Έχουμε την τύχη να είμαστε παρόντες σήμερα που γράφεται ιστορία. Και απαντώ και στον κύριο Ντεγκράφ. Δεν είναι ούτε πρώτη φορά, ούτε η τελευταία φορά που εσείς ε, βρεθήκατε στη λάθος πλευρά της ιστορίας. Χάσατε το ραντεβού σας. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τα μεγάλα προβλήματα της ανθρωπότητας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε και πρέπει να είμαστε περήφανοι για αυτό που πετυχαίνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόρσοκ, ε, πρόεδρο του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμε Γενική Γραμματέα, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και την εκτίμησή μου για, την, για τον ηγετικό ρόλο που διαδραμάτισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών στις, αυτές, στις κοινές προσπάθειες ε, να συμφωνήσουμε σε μια φιλόδοξη συμφωνία των Παρισιών και να σας ευχαριστήσω και για τις δεκαετίες υπηρεσίες σας προς τη διεθνή κοινότητα από τη θέση του Γενικού Γραμματέου των Ηνωμένων Αθηνών. Σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά διατρανώνει και πάλι την προσήλωσή της σε συνεχείς δράσεις για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέβαλαν και τους ευχαριστώ για την συνεργασία που είχαμε και ευχαριστώ θερμά και την Πρόεδρο Σεγκολένου Αγκιάρ για την αποφασιστικότητα και την προσπάθειά της ε, να επισπεύσει την κύρωση της Συμφωνίας των Παρισίων. Γιατί αυτή η δέσμευση αφορά την αξιοπιστία μας, την ευθύνη μας και το ρόλο που διαδραματίζουμε στο παγκόσμιο προσκήνιο. Γιατί εργαστήκαμε εργοδός στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία χρόνια για να διαμορφώσουμε τη νέα συμφωνία κατά των κλιματικών αλλαγών που διαμορφώθηκε και πήρε την τελική της μορφή στο Παρίσι. Και μάλιστα ε, στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης ε, Παρασκευής φάνηκε η υποστήριξη των κρατών μελών υπέρ της κύρωσης της Συμφωνίας των Παρισίων εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα το Συμβούλιο επίσημα θα ε, υιοθετήσει αυτή την απόφαση. Και μάλιστα από σήμερα θα ξεκινήσουμε να εφαρμόζουμε και εμπράκτος αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κότσο. Ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία της ψηφοφορίας και θα δώσω το λόγο πρώτα στον εισηγητή και πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος, κύριο Τζοβάνι Λαβία. Κύριε Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, συνάδελφοι, ε, κυρίες και κύριοι, ως πρόεδρος ε, της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος και εισηγητής θα ήθελα με ιδιαίτερη περηφάνεια να στήσω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει αμέριστα την κύρωση εκ μέρους Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Συμφωνία των Παρισιών. Πριν από 20 περίπου χρόνια το πρωτόκολλο του Κιώτο θαύτηκε από την Αμερικανική Γερουσία. Έκτοτε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστάτησε στι διεθνεί προσπάθειε να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή και εργάστηκε σκληρά για να στεφθεί με επιτυχία η Συμφωνία των Παρισίων. Η συμφωνία αυτή θα τεθεί σε ισχύ χάρη στην ε, απόφαση του οίκου των Ευρωπαίων πολιτών. Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή και είναι ο καρπός μιας τεράστιας συλλογική προσπάθειας των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των ε, μελών των Εθνικών Βουλών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κρατών μελών και των Προεδριών του Συμβουλίου. Θα ήθελα ιδιαίτερα να αναγνωρίσω και να πατήσω φόρο τιμή στον Επίτροπο Αρία Κανιέτε, με τον οποίο είχαμε στενέ και τακτικέ επαφέ καθ' όλη τη διάρκεια τη διαδικασία. Η σημερινή ψηφοφορία θα δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί τις υποσχέσεις που έχει κάνει. Ε, οφείλουμε και δυνάμεθα να, να ε, δώσουμε στις ερχόμενες γενιές έναν σταθερότερο κόσμο, πιο ευήμερο, υγιέστερο και πιο καθαρό πλανήτη. Σήμερα είμαστε κοντά σε αυτό το στόχο και σήμερα δυνάμεθα να το πραγματοποιήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί η ψηφοφορία τώρα για τη σύσταση για ε, απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τη Συμφωνία Πλαίσιο του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή και τη σχετική Συμφωνία των Παρισίων. Εξ Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Άρχεται η ονομαστική ψηφοφορία. haben alle Abgeordneten. Ψηφίσατε όλοι. Όντως, πέρας ψηφοφορίας. Εψήφισαν 679 βουλευτές, υπέρ 610. 610 to 38. Κατά 38 και 31 αποχές. Διαπιστώνω ότι το Κοινοβούλιο συμφώνησε με τη συμφωνία αυτή.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

Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμοι συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για τη συντριπτική πλειοψηφία αυτή και θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω όλους εκείνους τους συναδέλφους που εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά έτσι ώστε να ε, επιταχυθεί η διαδικασία αυτή η συνένεση. Θα ήθελα Εξ ονόματός σας να ευχαριστήσω και πάλι τον κύριο Μπαν Κιμούν, Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όχι μόνο για τη σημερινή του παρουσία, αλλά και για την εξαιρετική ηγεσία ε, στα Ηνωμένα Έθνη τα τελευταία δεκαετία. Για τις υπόλοιπες εβδομάδες και από εκεί και πέρα σας ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και στην προσωπική σας ε, ζωή. Όχι μόνο να έχετε πολλά καλά χρόνια μπροστά σας, αλλά να ξέρετε ότι τρέφουμε μεγάλο σεβασμό ε, στο πρόσωπό σας που ηγηθήκατε στην ΕΕ σε τέτοιους καιρούς δραματικούς και ταραγμένους. Ευχαριστούμε πολύ.